Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Οι προσκεκλημένοι μας είναι παρόντες. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας μας διάταξης για σήμερα. Φτάνουμε λοιπόν στο το τελευταίο σημείο για το οποίο θα έχουμε τη τιμή να ακούσουμε τρεις προσκεκλημένους. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις της TTIP για την συμφωνία δηλαδή για το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, από κοινού με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, που ασχολείται επίσης με το θέμα. Συνάδελφε ε, Λάγκ ε, συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, έχουμε εδώ να επικεντρωθούμε στις βασικές μας ανησυχίες, δηλαδή τις νητικές επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως στις λιγότερο προηγμένες χώρες. Η αντίκτυπο του TTIP ξεπερνά τις διμερείς μας σχέσεις στο βαθμό που αυτή η συμφωνία θα επανακαθορίσει τους κανόνες του παγκοσμίου εμπορίου και θα θεσπίσει και νέες μορφές. Ε, η Επιτροπή μα έχει ήδη πάρει θέση όσον αφορά τι διαπραγματεύσει μέσω ενός ψηφίσματος την περασμένη χρονιά, όπου ζητήσαμε από την Κομισιόν να ζητήσει ανεξάρτητη ανάλυση των επιπτώσεων του TTIP στι αναπτυσσόμενε χώρες, καθώ και σε σχέση με του στόχου ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Στην απάντησή τη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου μα, η Κομισιόν μα ε, διαβεβαίωσε ότι το TTIP θα ε, έχει τέτοια μορφή που θα είναι θετικό για τους άλλους μας εμπορικούς εταίρους και ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα θέλαμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι για αυτή την τη τύπη και είμαστε και πολύ περίεργοι να ακούσουμε την Επίτροπο, κυρία Επίτροπε, όσον αφορά τις προσωρινές, ε, τα προσωρινά πορίσματα της ε, μελέτης αντικτύπου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Με χαρά λοιπόν υποδέχομαι τους τρεις μας προσκεκλημένους, την κυρία Σεσίλια Μάρστρομ, Ευρωπαϊκή Επίτροπο Αρμόδια για το Εμπόριο, τον κύριο ε, Ιωαννού Νασουνού, υπό των χωρών ΑΚΕ και την κυρία Εβίτα Σμίγκ ε, στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας. Ε, θα σας καλέσω λοιπόν να πάρετε το λόγο και να, μιλ... και να κάνετε τις εισηγήσεις σα για 10 λεπτά. Ε, ε, στη συνέχεια θα ζητήσω από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που είναι εδώ παρόντες να ε, υποβάλουν ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις τους. Ε, πριν να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μα θα ήθελα να δώσω το λόγο προ... στον συνάδελφο Λάγκε που όχι μόνο είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, αλλά είναι και εισηγητής για το TTIP. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Πονγκά. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχουμε την κοινή συνεδρίαση σήμερα και μπορώ να προεδρεύσω μαζί με τον συνάδελφο πρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Όπως είπατε, κύριε Πόγκα, στις 8 Ιουλίου του 2015 με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο το ψήφισμα για το TTIP που αποτελεί και ένα μπούσουλα ε, τον ήρμο για την ε, τελική θέση του Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν καλό που και σε αυτό το ψήφισμα έχουν μπει πολλά στοιχεία που πρότεινε η Επιτροπή σας και που διατρανώσαμε ότι με τη συμφωνία αυτή θέλουμε να ε, ρυθμίσουμε τις εμπορικές ροές έτσι ώστε να είναι ελεύθερες αλλά και δίκαιες και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες των αναπτυσσόμενων χωρών και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να τις βοηθήσουμε και να τις λάβουμε υπόψη μας. Στο ψήφισμα λοιπόν της 8ης Ιουλίου του 2015 διατρανώσαμε ότι το TTIP το θεωρούμε εφαλτήριο ως ε, λοιπόν για μελλοντικές ε, συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ και όχι για διμερή μπλοκ που θα σχηματιστούν. Και ε, δεν ε, αμφισβητείται λοιπόν έτσι ούτε το θέμα της ΔΟΧΑ ούτε των υπολείπων συμφωνιών του ΠΟΕ. Την περασμένη εβδομάδα στην μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση στην Ισομερή με τις χώρες ΑΚΕ το ξαναείπαμε. Οι μεγάλες περιφερειακές συμφωνίες μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα και ευεργετήματα για τις μικρές χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες, βεβαίως εφόσον υπάρχει το σωστό πλαίσιο και οι σωστές προϋποθέσεις πάντα. Άρα και σήμερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είτε είναι αυτό το ζήτημα της πρόσβασης στο διμερή χώρο εμπορίου, είτε πρόκειται για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ή τη διάνοιξη σε τρίτες χώρες, ένα σωρό τέτοια θέματα. Ή να ασχοληθούμε με τις ρυθμίσεις για τις χώρες προέλευσης έτσι ώστε να μην παραγωνιστούν οι τρίτες ε, χώρες. Τώρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή του TTIP, ούτε είμαι βέβαιος ε, ότι θα δει το φως της δημοσιότητας το TTIP και θα γεννηθεί έτσι, στο προσεχές μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οφείλουμε να προβληματιστούμε και να δούμε τις δυνητικές συνέπειες σε τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, κατέθεσε ένα Sustainable Impact Assessment, τη μελέτη αντικτύπου, ε, τη βιώσιμη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη θέση των χωρών με χαμηλό εισόδημα ότι θα πρέπει να έχουν μια αύξηση του ΑΕΠ τους, έστω και μικρή. Αυτά. Ε, λοιπόν, είναι ωραίο και καλό που μας προβληματίζει αυτό, το θέμα σήμερα και με χαρά προχωρούμε σε αυτή την ακρόαση. Με χαρά θα ακούσω και τους προσκεκλημένους ομιλητές. Λοιπόν, αρχίζουμε. Très bien, merci, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πίτροπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Πόγκα, Πρόεδρε Λάγκε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ και τις δύο τις επιτροπές που διοργανώσατε αυτή τη συζήτηση. Είναι σωστό και ωφέλιμο και είναι σημαντικό όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και γιατί πολλοί πολίτε θέτουν αυτά τα ερωτήματα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εστιάζεται μόνο στο να αποφέρει οικονομικά πλανεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή την άποψη. Φυσικά, η εμπορική πολιτική σημαίνει δημιουργία ευκαιριών, δυνατότητε για ανάπτυξη και επενδύσει για του εργαζόμενου, του καταναλωτέ και του επιχειρηματίε μα. Πρέπει να υπερασπίσουμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντά του γιατί κανεί άλλο δεν θα το κάνει αυτό. Όμω είναι πολύ ευρύτερη υπόθεση. Είμαστε μια ένωση αξιών και συμφερόντων και είμαστε ένωση Δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε μια ένωση που επιμένει για την ε, προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, αλλά και είμαστε και μια ένωση που στηρίζει την ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών. Και αυτό είναι μια πολιτική που υποστηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους πολυσυμπολίτες μα. Το να μιλάμε λοιπόν για την ε, διατλαντική συμφωνία επενδύσεων και εταιρική σχέση και πώ επηρεάζει τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι διόλου παράξενο να το ρωτά κανεί αυτό. Καταρχά, γιατί η κλίμακα αυτή τη συμφωνία είναι πολύ μεγάλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ μαζί συναποτελούν το 50% τη παγκόσμια οικονομία, 40% των επενδυτικών αποθεμάτων και 30% του εμπορίου ε, και είμαστε εξαγωγικοί προορισμοί για τι 43 χώρε με με τα χαμηλότερα εισοδήματα ε, και θέλουμε να ξεπεράσουμε τα εμπορικά ζητήματα αλλά και τις πιο προηγμένες εμπορικές μας συμφωνίες. Θέλουμε να εξετάσουμε κανόνες και κανονισμούς που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα της ΣΥΤΙΠ θα επηρεάσει τον κόσμο αλλά και φυσικά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και το θέμα είναι πώς θα τις επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες εφόσον η Ένωση και η συνεργαστούν στενά στενότερα. Αυτό το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και για τις τρίτες χώρες εν γέννη. Και με χαρά μπορώ να σας πω ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει αρνητικό αντίκτυπος, αν και ακόμα ξεκολουθούμε να επαγρυπνούμε. Όλες οι μεγάλες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στο θέμα αυτό μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το TTIP θα είναι ωφέλιμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το πόρισμα των μελετών που κάναμε εμεί στην Κομισιόν, αλλά και εκτό και αντιστοιχεί και στα πορίσματα διαφορών εθνικών μελετών που έγιναν, α πούμε, στι κάτω χώρε. Γιατί το σημείο εκκίνηση είναι το βασικό στοιχείο για την παγκόσμια οικονομία. Όταν η Ένωση και η ΕΠΑ αναπτυχθούν από πλευρά τη οικονομία, αυτό σημαίνει αύξηση τη ζήτηση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και το αντίστροφο ισχύει βέβαια και το έδαμε μετά από την οικονομική κρίση η TTIP, καθιστώντα τι οικονομίε μα ισχυρότερε, θα ε, αναδείξει τη θετική πτυχή που θα, αυτό θα φανεί έμεσα γιατί όταν αναπτυσσόμαστε εμείς εισάγουμε περισσότερο και αυτό επηρεάζει θετικά τις αναπτυσσόμενες χώρες και έμεσα γιατί οι πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κομμάτια της λυσίδα προμηθειών προς τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ε, κάθε... Ε, κάθε ε, εκατομμύριο ευρώ, ε, δισεκατομμύριο συγγνώμη, ευρώ που επενδύουμε σημαίνει στήριξη σε 8.500 ε, ε, σε, σε 800.000 μάλλον θέσεις απασχόλησης παγκοσμίω, Βραζιλία, Ινδία κτλ. Η TTIP λοιπόν άρα δεν θα σήμαινε περισσότερο εμπόριο και άρα οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς θα είχαν πλεονεκτήματα απέναντι στι ε, εξαγωγέ των αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με τι μελέτε, όχι, γιατί οι αναπτυσσόμενε χώρε στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική ειδικεύονται σε πολύ διαφορετικά προϊόντα και από ότι οι Ευρωπαίοι κατά παραγωγή. Και αυτό είναι προφανέ γιατί η προστέμενη αξία από τις εξαγωγές σήμερα ε, σε προϊόντα δεν ανταγωνίζονται ε, τα προϊόντα της Αφρικής, ας πούμε, ε, και ούτε τα φαντουργικά προϊόντα που κατασκευάζονται πούμε, στο Μπαγκλαντές στην Ινδία ανταγωνίζονται τα δικά μας εδώ. Αυτό δεν... Όμως, αν αφαιρέσουμε τους δασμούς λοιπόν θα ωφεληθούμε και εμείς αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος και θα, ελάχιστα θα επηρεάσει τους υπόλοιπους. Η DTP έχει να κάνει και με τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο. Δηλαδή πώς θα είναι συμβατές οι απαιτήσει και οι προποθέσει δοκιμών για τα προϊόντα και αυτό δεν θα πρέπει να το αποθετήσει το τρίτα μέρη σε μειονεκτική θέση γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε προτιμήσεις στα προϊόντα της Ευρώπης ή του, των ΗΠΑ. Μάλιστα, θα αποτελέσει Τι τη βάση για τις μελλοντικούς παγκόσμιους κανόνες εμπορίου. Και επίσης η TTIP που περιλαμβάνει καθολικές διαστάσεις, ε, ε, περιλαμβάνει διάφορες διευκολύνσεις για τα τελωνία και το εμπόριο, πράγμα που θα, διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον τομέα των ρυθμιστικών φραγμών, ε, τα τρίτα μέρη μπορεί να ωφεληθούν άμεσα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ, ΕΕ, αν συμφωνήσουν σε κοινέ προσεγγίσεις, ας πούμε, για την αμοιβή αναγνώριση για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στα αυτοκίνητα, τα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτού τι προδιαγραφέ θα κυκλοφορούν και στι δύο αγορέ. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν δύο διαφορετικέ γραμμέ παραγωγή και αυτό σημαίνει ευκολότερη συμμόρφωση προ του κανόνε και τι προδιαγραφέ. Τέλο, Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το δεν συμβαίνει απομονωμένα. Συνεχίζουμε και τη δουλειά μα που, κάνουμε εδώ και καιρό για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των προϊόντων των τρίτων χωρών στι αγορέ μα. Ολοκληρώνουμε συμφωνίε με τη Λατινική Αμερική, αλλά η σχετική συμφωνία με το Μερκοσούρ. Διαπραγματευόμαστε για τον εξυγχρονισμό των εμπορικών εμπορικών συμφωνιών με το Μεξικό και τη Χίλη. Έχουμε κάνει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στι ε, ε, συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση. Πριν από λίγε μέρε ήμουν στην Ποτσουάνα και υπογράψαμε εκεί τη συμφωνία ΣΑΝΤΕΚ και στην Ανατολική Αφρική θα, θα, θα ε, υπογράψουμε σε λίγο καιρό την συμφωνία ΕΑΚ. Περαιτέρω δηλαδή άνοιγμα των αγορών μα για αυτέ τι χώρε. Με ασύμετρο τρόπο. Οι υπόλοιπε αφρικανικές χώρες έχουν δασμολόγητη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές ούτω ή άλλω. Τώρα, όλα τα μέλη του ΠΟΕ, οι 162 χώρε, ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενε χώρε, έχουν χρυσή ευκαιρία για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του εμπορίου του με τον υπόλοιπο κόσμο, κυρώνοντα τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Διότι αν υπάρχει στα σύνορα, ε, προσβάλλουν τις δυνατότητες των χωρών αυτών να εξάγουν ας πούμε, οι τελωνικές ε, διατυπώσεις ε, σημαίνουν πέντε περίπου έγγραφα ε, και 700 ευρώ κόστος ανά κοντέινερ. Στην υποσαχάρια Αφρική 35 μέρες παίρνει εξαγωγή, 45 μέρες η εισαγωγή και κοστίζει 1.300 ευρώ στην εξαγωγή και 1.500 ευρώ στην εισαγωγή το κάθε κοντέινερ. Και να σας πω στην Αιθιοπία ότι οι δασμοί διπλασιάστηκαν το τελευταίο χρόνο ε, και έφτασαν το 51%. Πολλά έχουμε να κερδίσουμε αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, και αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την TTIP. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το μονοπάτι οικονομικής μεταρρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως TTIP. Αυτά είναι τα πορίσματα λοιπόν των μελετών που έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Φυσικά ε, ξεκολουθούμε να εξετάζουμε το θέμα με πολύ πολύ φροντίδα και προσοχή και μελετούμε και την, ε, τον ευρύτερο αντίκτυπο όλων αυτών. Έχουμε δημοσιεύσει μια πρώτη έκθεση, θα δημοσιευθεί και μια επόμενη τέλη Ιουλίου και μια τελική έκθεση θα έχουμε στα τέλη του έτους. Οπότε σας καλούμε να σχολιάσετε το σχέδιο το οποίο μόλις δημοσιεύτηκε και θα το συζητήσουμε εξάλλου και σήμερα. Είναι πολύ επίκαιρη η σημερινή μα συζήτηση και φυσικά προσβλέπω στι ερωτήσει και τα σχόλιά σα, ε, με τα οποία μπορούμε να συμπληρώσουμε το τελευταίο κομμάτι τη έκθεση αντικτύπου μα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που με καλέσατε και ε, προσβλέπω στην υποψηνή συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την εισήγησή σα αμέσω θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νασουνού για 10 λεπτά επίση. Παρακαλώ. Merci. Euh. Σας ευχαριστώ, κύριε Συμπρόεδρε. Εξ ονόματος ε, των χωρών ΑΚΕ, σας ε, ευχαριστούμε που μας ε, ζητήσατε να συμμετάσχουμε και να συμβάλλουμε σε αυτή την συζήτηση. Ε, και κατά το παρελθόν ε, είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις ε, με την Επίτροπο. Έχουμε άλλωστε άπαξ του έτους συνάντηση ε, στην ε, ε, Υπουργική Επιτροπή Εμπορίου στο Κοτονού που μας δίνει την δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα και επίσης να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να ενδυναμώσουν την εταιρική μας σχέση. Ακούσαμε όσα είπε και σήμερα η Επίτροπος που ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις που έχουμε μέχρι τώρα λάβει ε, στους προβληματισμούς που έχουμε εκφράσει. Ωστόσο προβληματιζόμαστε ακόμα, γιατί όπως είπε και ο Συμπρόεδρος, ε, έχουμε πάλι ακόμα την εντύπωση ότι ένα μεγάλο τμήμα της οικονομικής ανάλυσης ε, βασίζεται σε υποθέσεις. Άλλωστε έτσι λειτουργεί η οικονομική επιστήμη. Σημαντικό είναι όμως να μάθουμε εάν ε, οι ε, συνθήκες που, και οι προϋποθέσεις ε, ισχύουν έτσι ώστε τα σενάρια να είναι πιθανά. Η ανάλυση έτσι όπως έχει γίνει στα διάφορα, στις διάφορες μελέτες είναι στατική. Στατική ενώ σε επίπεδο ΑΚΕ υπογράφουμε εταιρικές συμφωνίες, σχέσεις, συμφωνίες εταιρικών σχέσεων δηλαδή, που θα μας δώσουν την δυνατότητα να αναδιαρθώσουμε πλήρως τις οικονομίες μας. Όταν ακούμε λοιπόν μια ανάλυση που λέει ότι ναι, η παραγωγή πρώτων υλών στις χώρες ΑΚΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική διάρθρωση της Αμερικής ε, ή της, ε, των χωρών της Ευρώπης, ε, τότε κατανοούμε ότι η δυναμική δεν είναι σωστή. Και άλλωστε εμείς δουλεύουμε ε, προς ε, την κατεύθυνση αυτή ε, βλέπουμε ότι οι χώρες ΑΚΕ μπορούν να είναι και χώρες παραγωγή και χώρες που εξάγουν τελικό προϊόν. Και όταν έχουν φτάσει στο επίπεδο που τους επιτρέπει να σέβονται τις διεθνείς αρχές, τότε μπαίνουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν δεν προωθείται μέχρι τέλους η, η υπόθεση εργασίας. Βεβαίω συμφωνούμε ότι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ε, η υποσυζήτηση συμφωνία μπορεί να παρουσιάσει και θετικά στοιχεία για τις χώρες ΑΚΕ. Εάν ε, η ευρωπαϊκή οικονομία και αν και η αμερικανική οικονομία ανακάμψουν, τότε αυτό είναι πολύ θετικό εάν οι τιμές εξαγωγής αυξηθούν με την οικονομική ανάκαμψη και αυτό θα μπορεί να έχει ε, ικανό αντίκτυπο στις χώρες μας. Αλλά για την ώρα έχουμε μια στατική αντιμετώπιση της ε, ε, οικονομίας γιατί εμείς εξακολουθούμε να είμαστε εξαγωγής πρώτων υλών. τα, οι επιδοτήσεις επίσης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Απογοητευτήκαμε λίγο γιατί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου δεν καταφέραμε ε, να ε, προωθήσουμε τα δικά μας αιτήματα. Πράγμα που μας οδηγεί στην ε, ερώτηση Θέλουμε μήπως να φύγουμε από το διμερές ε, επίπεδο και από τη διμερή, σχέση και ίσως να βολέψουμε ας πούμε τα πράγματά μας, ε, τα δικά μας με συμφωνίες μεταξύ φίλων. Ε, θα ήταν κατανοητή μια τέτοια κίνηση, αλλά όπως είπε και η ίδια η Επίτροπος, η συμφωνία η οποία θα επιτευχθεί ε, από τις μεγάλες οντότητες οπωσδήποτε θα έχει ε, και επίπτωση και στις ε, διεθνικές συμφωνίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο και αντίστοιχα να αυξήσουμε το θετικό αντίκτυπο τέτοιων κινήσεων. Δεν θα επανέλθουμε στο θέμα των προτιμήσεων γιατί μπορεί και η μία πλευρά να έχει κάποιες ε, μελέτες που αποδεικνύουν το α, αλλά και εμείς μπορούμε να ε, βγάλουμε μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν το αντίθετό του. Επίσης, όσον αφορά το ρυθμιστικό επίπεδο, μέχρι τώρα κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Σύσταση για τις ε, ρυθμίσεις εξελίσσεται, ε, πρέπει να δίνεται κάποια δυνατότητα χρονική και άλλη στις ε, χώρες μας για να ε, προσαρμοστούμε. Εδώ όμως αυτό που κινδυνεύει να συμβεί είναι να μείνουμε λίγο στην άκρη και να μην μας δοθεί η ίδια δυναμική. Ας πούμε, έχουμε μπροστά μας σοκολατάκια. Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα ενός παραγωγού στην Γκάνα και που ε, φτιάχνει σοκολάτες και τις εξάγει ε, και εξάγει στην ευρωπαϊκή ε, αγορά υποχρεούμενος να σεβαστεί ορισμένους κανόνες. Εάν υπάρξει μια συμφωνία επί των νέων κανόνων με την αμερικανική πλευρά ας πούμε και επομένως με ένα ρυθμιστικό ή νομοθετικό ε, επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με τις εξαγωγές από την Κάνα, τότε και λαμβάνοντα υπόψη τι μεγάλε θυσίε που απαιτεί η Ευρώπη από του παραγωγού τη Γκάνα, τότε οπωσδήποτε θα στραφούν οι παραγωγοί της Γκάνα προ ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, και καταλαβαίνετε ποιο μπορεί να είναι ο αντίκτυπο, λαμβάνοντα υπόψη και τις οικονομίες κλίμακο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να καταλάβουν όλοι ότι αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι μια δυναμική και δυναμικά εξελισσόμενη και κινούμενη οικονομία οικονομία η οποία να είναι σε θέση να παράγει πλέον μεταποιημένα τελικά προϊόντα υψηλότερης ε, αξίας. Θέλουμε όμως από την άλλη πλευρά να έχουμε και όλες τις προσήκουσες και απαραίτητες ε, ε, πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ε, μια σωστή ανάλυση. Ναι, έχουμε ανταλλαγές, αλλά πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για περισσότερες πληροφορίες από πλευράς των εταίρων μας. Από την δική μας πλευρά εμείς λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε πιο ενδελεχή μελέτη ε, επί τη βάση συγκεκριμένων ε, στοιχείων. Έχουμε κάνει και τώρα κάποιες αναλύσεις ε, επιβάσεων βάσεων όμως και επί στοιχείων ιδιαίτερως υποθετικών. Σας έδωσα ένα παράδειγμα για τη σοκολάτα, αλλά αντίστοιχα παραδείγματα μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε τη φιλοδοξία καθόλου να, να δημιουργήσουμε εμπλοκές. Θέλουμε να παραμείνουμε θετικοί και θέλουμε με θετικό πρόσημο να συνεχίσουν οι σχέσεις μας. Αυτά, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, ήθελα να σας πω. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το μέλλον και τις μελλοντικέ μας κινήσεις και είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες βεβαίως. Σας ευχαριστώ, κύριε Γνασουνού. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Εβίτα Σμιτ, καθηγήτρια, την οποία ε, είχαμε τη χαρά να ακούσουμε και την προηγούμενη χρονιά. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και δεν είμαι καθηγήτρια, μια απλή διδάκτορη είμαι. Ε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω και τις δικές μου απόψεις για τις δυνητικές συνέπειες του TTIP στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Συμφωνώ με τα όσα ήδη υπόθηκαν, με ορισμένα διαφωνώ. Ε, για να συνεισφέρουμε σε μια ζωηρή συζήτηση θα ήθελα να διαρθρώσω ε, την ομιλία μου σε έξι σημεία παραδοχές και συστάσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη να ελαχιστοποιήσει τις ανετικές συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει. Αυτό είναι το θετικό. Δεύτερη ε, θετική συνέπεια, ε, ε, τα πρότυπα θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν. Τρίτον, η TTIP θα πρέπει να προσέξουμε να μην οδηγήσει και περαιτέρω περιοθεοποίηση της μικρός χώρες. Η ΕΠΑΣ, η ΣΟΕΣ, ε, θα πρέπει να βοηθήσουν να μετριαστεί αυτό το ενδεχόμενο, πράγμα που δεν είναι πάρα πολύ πιθανό. Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθάει τις μικρές χώρες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά και έκτον, ε, η ε, στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, εάν εφαρμοστούν, αυτό θα σημάνει και καλύτερη μοίρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει την ευθύνη να ελαχιστοποιήσει τις ανετικές συνέπειες. Έχει ευθύνη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό απορρέει από την πολιτική συνοχή τη συνεκτική πολιτική στην οποία υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν πέρσι. Ο βασικός κίνδυνος εδώ για το εμπόριο προέρχεται από ε, την παράκαμψη του εμπορίου, ιδιαίτερα σε τομεί που είναι υψηλή ακόμα οι δασμοί, όπως είναι τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα κλωσοεφαντουργικά και τα υποδήματα κυρίω. Και η κυρία Μάλμστρομ είπε φυσικά και έχει δίκιο, δεν χωράει καμία αμφιβολία περί αυτού, ότι οι δομές παραγωγής και εξαγωγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών διαφέρουν πολύ σε σχέση με εκείνες των φτωχών κρατών. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από εκεί. Παραμένει όμως ε, το ενδεχόμενο σε ειδικά προϊόντα να υπάρξει αυτή η στρέβλωση και ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έκβαση θα έχει το TTIP, αλλά δεν αποκλείεται να πλήξει ορισμένα προϊόντα και να γίνουν κάποιες παρακάμψεις στο εμπόριο εις βάρος των φτωχών κρατών. Θετικά επίσης αναφέρθηκαν για τις χώρες που συμπεριλαμβάνονται ε, στην αλυσίδα παραγωγής αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πολιτειών. Αυτό αφορά τις μάλλον πιο ανεπτυγμένες χώρες. και όχι τις λιγότερο ανεπτυγμένες, γιατί διαφέρει η δομή των εξαγωγών τους. Λοιπόν, υπάρχουν συστάσεις. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, από διάφορες αφετηρίες για να αποτρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες. Πρώτον, υπάρχουν οι κανόνες για τη χώρα προέλευσης. Εδώ δεν θα πρέπει ε, να σορευτούν πολλοί εταίροι ε, με συμφωνίες FTA, ελευθέρων συναλλαγών ή ε, προτιμήσεων. ορισμένοι λέγουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου κανόνες για τη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, χαλαροί οι ασήμαντη, αυτό δεν θα ήταν ε, προ όφελο των ε, φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά το πιο ανεκτημένων, Βλέπε Κίνα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός ε, στο TTIP για να υπάρχουν περιορισμοί, μάλλον να, να παλινθούν κάπως ενετικέ συνέπειες. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτείες θα μπορούσαν μονομερός να μετριάσουν τα GSP. του στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Which are sectors, countries and products concerned, and it would be possible to adapt the respective GSPs. Second assumption, I think I don't have to... Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, συγγνώμη. Ε, ε, το TTIP θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία ρήτρα ειδική που να επεκτείνει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πολιτειών σε αμοιβαία αναγνώριση ή ε, κάτι αντίστοιχο που μπορεί να επεκταθεί σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε το κάθε πλεονέκτημα ε, στον τομέα αυτό να είναι και προς όφελος των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών. Τρίτη παραδοχή. σε πολύ μικρές αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει αυτές να βοηθηθούν να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Ήδη από σήμερα είναι περιθωριοποιημένες, Η υποσαχάρη Αφρική στις παγκόσμιες εξαγωγές συμμετέχει μόνο κατά το 1,7% και 2% μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό ε, δεν... Δεν είναι αυτό όμως ε, το φταίξιμο του TTIP ή η διαφορετική μεταχείριση στον ΠΟΕ. Παρόλο που έχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την κατάσταση αυτή. Εάν το TPP και το TTIP, αυτές οι μεγάλες περιφερειακές ε, συμφωνίες θέλουν να επιτύχουν, θα πρέπει ε, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κέντρα στην παγκόσμια οικονομία και αυτό θα σήμαινε ότι περιθωριοποιούνται ακόμα περισσότερο οι φτωχέ μη ανεπτυγμένες χώρες, επιβαρύνονται από τεχνικές προδιαγραφές που δεν μπορούν να καλύψουν και δεν μπορούν να συμμετέχουν και όλα στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι θα μπορούσαν να εποφεληθούν από την ανάπτυξη που θα έρθει στις χώρες Αλλά αυτές οι παραδοχές είναι πάρα πολύ γενικές και αν υπάρξουν βεργετήματα θα είναι τις προ, προς τις πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες και όχι τις πιο φτωχές. Βλέπω ότι φεύγει και ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Ένα σημείο μόνο. Αν οι μέγα περιφέρειες λοιπόν μάλλον θέλουν να είναι επιτυχείς ε, και να μετριαστεί αυτή η περιθωριοποίηση των μικρών ανεπτυσσόμενων χωρών, πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Και οι BRICS, ε, οι αναδυόμενες μεγάλες οικονομίες, δεν συμμετέχουν στις μέγα περιφέρειες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο για να συμμετέχουν περισσότερο στον ΠΟΕΣ, το διεθνές στερέωμα, γιατί φυσικά φοβούνται για τις ε, επιπτώσεις που θα υποστούν οι μικρές χώρες. Τέταρτη παραγωγή, παραδοχή, συγγνώμη. Η ΕΠΑΣ, η συμφωνίες οικονομικής ε, εταιρική σχέσης, ΣΟΕΣ, ε, καλύπτουν διάφορους τομείς, τεχνικές προδιαγραφές, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων κτλ. Θα μπορούσε ε, αυτό να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να συμμορφωθούν με υψηλότερα στάνταρ. Ωστόσο, αυτές οι ρήτρες που μπορεί να είναι χρήσιμες συμπεριλαμβάνονται στις ΣΟΕΣ, στο στις διατάξεις λεγόμενες ΠΟΕ που δεν αφορά κυρίως στις αφρικανικές χώρες. Στην Καραϊβική οι ΣΟΕΣ είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν γιατί είναι θετικές διατάξεις ευνοϊκές, μη δεσμευτικέ όμως, προαιρετικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά να προωθηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Οπότε έχω τις επιφυλάξεις μου κατά πόσο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πέμπτη παραδοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει για τη βοήθεια με αντάλλαγμα το εμπόριο, να κάνει μια λεπτομερή ανάλυση αναχώρα. Είπατε ότι αυτό χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις TTIP και έχουμε την πραγματική συμφωνία. Από εκεί και πέρα μόνο μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση και οι επιπτώσεις θα είναι πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά για να βελτιώσουν και τις ποιοτικέ του υποδομές και τη συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο. Τελευταία παραδοχή, η εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει πάρα πολύ επίση. Όλες οι εμπορικέ συμφωνίες, όσο καλές και να είναι, είναι μόνο εμπορικέ συμφωνίες. Αυτό το είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες και στο εξωτερικό και στις διεθνείς δομές και στο εσωτερικό υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μεμονωμένων χωρών στις εξαγωγικές αγορές. Η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης του 2015 αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα ζητήματα. Υπάρχει στόχος 17 που λέει ότι δεσμευόμαστε για διεθνούς κανόνες, διεθνείς κανόνες για ένα σύστημα χωρίς διακρίσεις πολυμερές στα πλαίσια του ΠΟΕ. Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να δούμε τι περιλαμβάνουν αυτοί οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ποια είναι η εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από το TTIP. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία μου. Θα ήθελα εξ ονόματος όλων να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους για τις παρεμβάσεις και θέλω τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση παρακαλώ να πάρουν το λόγο οι βουλευτές θα αρχίσουμε από την κυρία Μαρία Ρένα Σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις τρεις παρεμβάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερως διαφωτιστικές δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα γιατί έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πέντε ε, σημεία θέλω να θίξω. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Εδώ και 14 χρόνια ε, ο κύκλος της Ντόχα ε, στο, στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου έχει μπλοκαριστεί λόγω των κυρίως των απαιτήσεων των χωρών του Νότου πώς προωθούνται αυτές οι ε, διεκδικήσεις σε σχέση και με τις αξίες που έχει η Ευρώπη. Πώς λοιπόν σε μια συμφωνία όπως το TTIP ε, ε, προωθούνται αυτές οι διεκδικήσεις οι αντίστοιχες λοιπόν που είχαν οριστεί από τις, και είχαν αναφερθεί από τις χώρες του Νότου στον Διεθνή Οργανισμό εμπορίου. Πώς η Ευρώπη ε, μπορεί και μπόρεσε να είναι η Ευρώπη των αξιών. Δεύτερη, δεύτερο σημείο. Κυρία Μάλστρομ, είπατε ότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, γεννούν ανάπτυξη. Μπορούμε πολύ να συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή Ίντε και θέλουμε πραγματικά να πιστέψουμε αυτή τη δήλωσή σας. Δυστυχώς όμως η ανάπτυξη αυτή δεν δημιουργεί ανάπτυξη για τους άλλους. Και επομένω, αν δούμε τα διάφορα, τις διάφορες στιγμές ανάπτυξης της Ευρώπης ε, δεν οδήγησαν απαραίτητα σε ανάπτυξη ε, της ε, ΛΕΧΑ και επομένως, της ΛΑΧΑ και επομένως κατά αυτή την έννοια οι ασφάλειες οι οποίες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν σε μια χώρα δεν οδήγησαν άμεσα στις ή στην ανάπτυξή τους. Επομένω, θα πρέπει να μα δείτε, να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην Αφρική, κυρίως όσον αφορά το μεταποιημένο προϊόν. Γιατί, ναι, ε, ε, ε, εάν αναπτυχθεί η Ευρώπη και χρειάζεται περισσότερη, ας πούμε, περισσότερο πετρόλαιο, ναι, θα αυξηθούν οι εξαγωγές πετρελαίου. Το ζήτημα όμως είναι αν αυτές οι χώρες θα αποκτήσουν την δυνατότητα να μεταποιούν και να εξάγουν μεταποιημένα τελικά προϊόντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κυρίως γιατί δεν είμαι βέβαιη ότι οι εμπορικές ε, συμφωνίες οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Ε, μπορώ να αναφερθώ και στις ε, συμφωνίες ελεύθερων ανταλλαγών με τις χώρες, Aid for Trade, με τις χώρες της Αφρικής, αλλά είδαμε ότι δεν έχουν προωθηθεί πάρα πολύ οι μεταποιητικές δραστηριότητες. Επομένως, αυτή η δήλωση ότι αύξη, ε, συγγνώμη, ανάπτυξη στην Ευρώπη ε, σημαίνει απαραίτητα και ε, ανάπτυξη στην Αφρική δεν ισχύει. Τρίτον, Ευρώπη αξιών. Συμφωνώ με σας. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά η Ευρώπη βλέπω ότι είναι έτοιμη ε, να υπογράψει συμφωνία με χώρες της Ανατολικής Αφρικής, μεταξύ των οποίων και το ε, ε, Μπουρούντι. Ενώ έχουμε το άρθρο 96 του, της Συμφωνίας Κοτονού που ρητά αναφέρει ότι το Μπουρούντι είναι χώρα η οποία σαφώς δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Ακούω ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ε, με την, ε, ε, ανταλλαγών, συγγνώμη, με την με τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής μεταξύ των οποίων και το Μπουρούντι. Νομίζω ότι είτε θα πρέπει να πούμε ότι εάν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κάνουμε δουλειά και δεν κάνουμε εμπόριο ή θα πούμε business as usual και τελείωσε. Επόμενο σημείο. Ο κύκλος της ε, Ντόχα ε, σκάλωσε κυρίως ε, στην γεωργία. Τώρα στη συμφωνία με τους Αμερικανούς αναφερόμαστε σε ένα τρόπο παραγωγής που είναι εντατικοποιημένη παραγωγή. Ε, τρόπος ε, παραγωγής ε, που έχει επικριθεί ιδιαιτέρως και όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και όσον αφορά και την διατροφική ασφάλεια και την διατροφική κυριαρχία. Επομένως, ένα μοντέλο σε αυτή τη συμφωνία TTIP τέτοιου είδους σημαίνει ότι, ότι δεν προωθούμε κάποιες άλλες μορφές ανάπτυξης οι οποίες στην Αφρική μπορούν καλύτερα να σεβαστούν τις αρχές Επόμενο σημείο. Γίνεται πολλή λόγος για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Αφρική. Όπως και στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο εμπόριο γίνεται ε, ε, εντός της περιφέρειας, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αφρική θα πρέπει επομένω να αναπτύξει τη δικιά της εσωτερική αγορά. Και σήμερα έχουμε την εντύπωση ότι και οι συμφωνίε TTIP και οι συμφωνίε που έχουμε με τις διάφορες περιφέρειες τη Αφρικής δεν σέβονται αυτήν την, την ιδέα της εσωτερικής περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. κυρίω το θέμα της ανάπτυξης μιας μεγάλης εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, Να κάνω μια διευκρίνηση. Έχω ακόμη 7 συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Βλέπετε όμως ότι το ρολόι γυρνάει. Θα σας ζητήσω λοιπόν να περιοριστείτε στα 3 λεπτά, ώστε να μπορέσουν μετά και οι καλεσμένοι μας να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι τελικά περί τίνος πρόκειται. Τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με εμβάσματα, να στέλνουμε λεφτά και να ε, ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε εμείς και να δημιουργήσουμε πλαίσια ε, που να μπορούν με κανόνες οι αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν μόνες τους ε, και να ευημερούν. Και το θέμα δεν είναι να μοιράζουν λεφτά που τους στέλνουν κάποιοι. Ε, η κατάρτιση εκπαίδευση και η μετακπαίδευση παίζει μεγάλο ρόλο και οι υποδομές βέβαια, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο είναι το aid for trade, δηλαδή να στέλνουμε βοήθεια για το εμπόριο, να καθόμαστε παραστάτες, να τους βοηθήσουμε, να βελτιώσουν τη διοίκησή τους, πώς μπορούν να λειτουργούν καλύτερα το δημόσιο και να κάνουν περισσότερα πράγματα για τους πολίτες που μπορεί άνδρες και γυναίκες. Και σήμερα με τις εξαγωγές ε, μπορούν να δημιουργηθούν εξαγωγικές επιχειρήσεις, ε, α, αυτοπασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικές. Με τις μεγάλες πολυεθνικές δεν είχαμε πάντα πολύ θετικέ εμπειρίες. Έρχονται, τα ρυθμίζουν όλα μόνοι τους, κανονίζουν, παίρνουν ό,τι θέλουν και χαίρεται. Ε, εδώ ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ευκαιρία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, για την ευελιξία της αυτοαπασχόλησης και η TTIP μας δίνει ένα τέτοιο πλαίσιο που ανοίγει νέε δυνατότητες για την εξάλληψη της γραφειοκρατίας ε, και την καταπολέμηση της διαφθοράς κυρίως. Στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε μέγα πρόβλημα με τη διαφθορά η οποία αποτρέπει πολλές δραστηριότητες και παραλύει. Οπότε θα πρέπει ε, ε, ο ανταγωνισμός να ξεφορτωθεί εκεί τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια, να απελευθερωθεί και αυτή είναι η μεγάλη αποστολή της Ευρώπης και της Αμερικής, γιατί ορισμένοι έχουν βολευτεί και πιέζουν τον κόσμο για φόρους, γιατί όταν είσαι μονοπόλιο και έχεις απέναντι το λαό, δεν μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει. Η Ευρώπη χρειάζεται ε, το θάρρος να προωθεί τις διεθνείς συμφωνίες και τη δίκαιη συνεργασία. Γι' αυτό χρειάζεται και διαφάνεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μείνατε στο χρόνο που σας έδωσα και τώρα το λόγο έχει συνάδελφος Ντέβα. Uh, um, Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι απλοϊκός άνθρωπος. Εάν βελτιώσουμε αμοιβαία τις προδιαγραφές μας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΕΠΑ, πράγμα που είναι το TTIP, να βελτιώσουμε τις διάφορες προδιαγραφές, τα υγειονομικά προϊόντα και ούτω καθεξής, προς τα πάνω, προς το πάνω οι προδιαγραφές, πώς αυτό θα γίνει συμβατό με τις αναπτυσσόμενε χώρες που κινούνται Πώς οι αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν ξαφνικά από το μηδέν θα πάνε στην τήρηση αυτών των εντυπωσιακά ψηλών προδιαγραφών που εμείς θα βάλουμε στο TTIP. Δεν τους κλείνουμε απ' έξω από τις αγορές μας. Όπως ε, στις αλληλευτικές συμφωνίες ας πούμε αποκλείουμε τις εισαγωγέ διαφόρων προϊόντων όπως οι γαρίδες ε, λόγω ακριβώς αυτών των υψηλών προδιαγραφών. Άλλα θέματα, κατεργασία φρούτων και λαχανικών. Εμείς όταν μιλάμε για προστιθέμενη αξία, στις χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πάρα πολύ ψηλέ ε, προδιαγραφές, πράγμα που μάλλον δεν θα μπορέσουν να κάνουν. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι αρκετά προβληματισμένος για το κατά πόσο οι διαπραγματευτές θα ασχοληθούν αποκλειστικά μόνο με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό αντίκτυπο. Νομίζω πως όλοι θέλουμε και στηρίζουμε την αρχή της σύγκλησης προς τα πάνω. Αν αυτή η αρχή δεν τηρηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το TTIP, οι περισσότεροι βουλευτές εδώ, σε αυτό το σώμα, δεν θα στηρίξουμε αυτήν την διαπραγμάτευση. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι θετικό για την ποιότητα είναι καλό για τους καταναλωτές της ΟΝΥΠΑ και για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι καλό για 800 εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, Όμως είναι προβληματικό και το είπε και η κυρία Σμίτη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι θα έχουν προβλήματα για να προσαρμοστούν στον ρυθμό αύξησης της ποιότητας δέχομαι ότι δεν μπορούμε να, λύσουμε στο, να ζητήσουμε από το εμπόριο να λύσει τέτοιου είδου προβλήματα. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο στην υπόθεση που εγκρίνεται αυτή η συμφωνία θα εξαρτηθούν λοιπόν όλα από τον τρόπο με τον οποίο θα συνοδευτούν αυτέ οι πολιτικέ. Τα μέσα λοιπόν αρκούν για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενε χώρε να προσαρμοστούν ε, στι ψηλότερε προδιαγραφέ για να μπορούν να εξάγουν προς την ε, Ένωση. Γιατί ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύψουν την διαφορά που ήδη υπάρχει, αν επιπλέον με τα ωφέλη της οικονομίας κλίμακας που θα γίνει μετά από την έναρξη ισχύω ενός τέτοιου συστήματος, η διαφορά, το χάσμα θα βαθύνει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε, πιστεύω, εξαιρετικά προσεκτικοί και επιπλέον εμείς είμαστε η Επιτροπή Ανάπτυξης. Η δική μας πρώτη αποστολή είναι λοιπόν να, που, να προσπαθήσουμε να εκριζωθεί η φτώχεια γι' αυτό και τονίζουμε τις συνοδευτικές πολιτικές. Είμαστε επίσης, επειδή θέλουμε να έχουμε συνοχή στις πολιτικές μας, χρειάζεται να, να τηρούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε προηγούμενες ε, σκέψει ε, όπως η τη Αντισαμπέμπα και τη Νέα Υόρκη για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξης. Δεν σημαίνει ότι επειδή το εμπόριο αναλαμβάνει περισσότερους κινδύνου στι αναπτυσσόμενες χώρε ότι, έχουμε, ότι είναι και λιγότερη φτωχή. Όχι. Δεν σημαίνει. Δεν συμβαίνει αυτό. Το εμπόριο το ίδιο από μόνο του δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα στο συνεπές εγχείρημα ε, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει το εμπόριο και η αναπτυξιακή πολιτική και κυρίως τα μέσα που μπορούν να κινητοποιήσουν αφρικανικές χώρες να προσεχθούν όλος ιδιαίτερος. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες μέσα σε αυτές τις αναλύσεις, ώστε να διευκρινίσουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε ω συνοδευτική πολιτική, όπως λέγεται. Και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σαφείς και συνεπείς σε αυτό. Και είναι ένα πραγματικό τεστ αντοχής όσον αφορά τη συνοχή, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Η Κομισιόν, λοιπόν, ως συλλογικό όργανο θα πρέπει να μας κοινοποιήσει αυτή τη νέα αταγική για να δούμε ποιος μπορεί να κάνει τα όσα δεν καταφέρει να κάνει το εμπόριο. Το εμπόριο από μόνο του δημιουργεί πλούτο, αλλά δεν σημαίνει ότι ε, λιγοστεύουν οι φτωχοί αυτό. Δεν θέλω να μαλώσω την κυρία Μάλστρομ για πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει κάποιος άλλος. Αλλά έχω να μαλώσω την Επιτροπή αν δεν μπορεί να μας παρουσιάσει μια συνεπή ε, γενική στρατηγική. Ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο θα πάρει τώρα η κυρία Λούλα Σάντσες. Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόγκα. Ερωτήσεις και σχόλια μου απευθύνονται στην Επίτροπο Μάλμστρομ. Εσείς ε, έχετε μια θέση μέσα στο έγγραφο εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη όπου υπερασπίζεστε την κοινωνική συλλογική ευθύνη ως τρόπο να ελέγξετε καλύτερα τις εταιρείε και ως εγγύηση και το λέτε ρητά ε, ως ε, τρόπο ελέγχου για το σεβασμό των εγχωρίων ε, νομοθεσιών και ο τι λέει ε, αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν άλλοι. Ε, φιλοσοφία, σε τι φιλοσοφία βασίζεται αυτά τα γενικά στάνταρ, γιατί όταν πρόκειται για την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών και για δημιουργία θέσπιση μάλλον σαφέστατων μηχανισμών με δυνατότητα επιβολής χειρώσεων, τα λέτε ξεκάθαρα. Όταν όμως θέλουμε, μιλάμε για έλεγχο των δράσεων των επιχειρήσεων εκτός Ένωσης ή σε οποιοδήποτε χώρο, στην ουσία επαφίεστε στη βούληση, στην καλή θέληση των ίδιων των εταιριών. Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και δεν θα λειτουργήσει οι πολίτες ε, γενικά του Νότου θα μπορούσαν κάτι να, σε κάτι να συμφωνήσουν αν υπήρχαν κάποια δεσμευτική, κάποια δεσμευτική όρη για τις επιχειρήσεις και να φέρομαι στην Ολομέλεια όπου είπαμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Ισπανική Inditex τις οποίες οι προμηθευτές ε, δρούσαν στο Μπαγκλαντές δεν θέλησε να αποζημιώσει τα θύματα ε, του ατυχήματος που συνέβη εκεί. Επίσης θέλω, θέλω να σας ρωτήσω ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε πως είναι συμβατή η TTIP με την εφαρμογή των, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί δεν υπάρχουν πουθενά, δεν αναφέρονται πουθενά στο TTIP. Άρα λοιπόν ε, τι θα κάνουμε, υπογράφουμε διάφορα ωραία πράγματα ε, για να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες, αλλά τελικά μένουν μόνο στα χαρτιά. Και να σας πω και ένα, ένα κάποιο προβληματισμό μου, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος Μαρία Ρένα, ότι είμαστε Ένωση Αξιών και Δημοκρατίας. Όμως δεν πάβουμε να είμαστε αυτό. Από τη στιγμή που στηρίζουμε κάποιες αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά χωρίς να είμαστε σε ένα παγκόσμιο φόρουμ και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη φωνή της πλειοψηφίας ε, του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η δημοκρατική συμφωνία, για να μην πούμε για τη διαφάνεια κτλ. Ξέρουμε ότι θέλετε να μπει αυτή η συμφωνία να εγκριθεί και να εγκριθεί και η ΣΕΤΑ. Πρόκειται όμως για μια τροπολογία που αλλάζει το νομοθετικό και δικαστικό σύστημα. Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό είναι ο τρόπο να εφαρμόζονται οι κανόνε σε διεθνέ επίπεδο, δηλαδή με τη βία. Μας λέτε... Μα λέτε ότι λείπει ο χρόνο, ότι πρέπει να κάνουμε γρήγορα, όμω η δημοκρατία παίρνει χρόνο. Και θα ήταν, νομίζω, ο καλύτερο τρόπο αυτό για τη θέσπιση διεθνών στάνταρ, γιατί τότε θα συμφωνούσαμε όλοι. Ευχαριστώ, η κυρία Χόιμπους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το πάνελ για τα όσα μας είπατε. Ε, καλά είπατε ότι είμαστε η Επιτροπή Ανάπτυξης εμείς και για νεωστή φορά θέλω να πω ότι η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική έχει προειδοποιήσει και για τις συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης και για το TTIP ότι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες θα υπονόμευαν την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική. Σας ερωτώ λοιπόν κυρία Επίτροπε, σε ποιο βαθμό λαμβάνονται αυτά υπόψη. Ε, αυτό το όργανο δεν είναι και ευκαταφρόνητο, δεν είναι καμιά επιτροπούλα. Είναι η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική. Έχει λόγο. Ε, και σε περίπτωση που εξαφανιστούν οι προτιμήσεις θα είναι εις βάρος του ισοζυγίου πληρωμών και τρεχουσών συναλλαγών των χωρών της Αφρικής. Αυτές είναι κάποιες προβλέψεις και προγνωστικά που δεν μπορούμε έτσι να τα παραγωνίσουμε ελαφρά την καρδία. Η κυρία Δόκτωρ Σμίγκ είπε ότι χρειαζόμαστε αναλύσεις πολύ συγκεκριμένες και ακριβείς έτσι ώστε να βρούμε ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες και να τις περιορίσουμε στο ελάχιστο. άρα εσείς υπολογίζετε ότι θα υπάρχουν, έτσι. Ε, οπότε πρέπει να συζητηθούν και αυτές κατά τη γνώμη μου και να τις ε, αξιολογήσουμε. Έχουμε ακούσει τις μεγάλες ανησυχίες των χωρών και τις ακούσαμε και σήμερα, αλλά και την περασμένη εβδομάδα στο Windhoek. Και βασική ανησυχία είναι αυτές οι προδιαγραφές. Αυτοί οι κανόνες και οι τιμές σε μια συμφωνία εμπορικών συναλλαγών μεταξύ δύο μεγάλων ε, εμπορικών εταίρων, Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι θα μείνουν εκτός νυμφώνος, γιατί δεν έχουν συζητήσει καν στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά τα πράγματα δεν οφείλουμε εμεί μόνο να τα λαμβάνουμε υπόψη, να, μάλλον να λαμβάνουμε απλώς γνώση, αλλά να τα λαμβάνουμε και υπόψη και να δούμε πώ θα προχωρούμε. Δεν μπορούμε εμεί να θέτουμε τι προδιαγραφέ για την υπόλοιπη υφήλιο. Αυτό δεν είναι μια συμπεριφορά πάρα πολύ... Ε, δέουσα και χωρίς αποκλεισμού στην ε, αναπτυξιακή μας πολιτική καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες στις χώρες αυτές να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να βοηθήσουμε να στηθεί μια παραγωγή, εν πάση περιπτώσει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε και ότι όταν παράγουμε σε αυτές τις χώρες και τις βγάζουμε από αυτό το ρόλο των αμυγός ε, εξαγωγικών χωρών, ορυκτών προϊόντων, <laughs> πρωτορελών, θα χάσουμε εμείς κάποιο μερίδιο, γιατί αυτοί εξάγουν την πρώτη ύλη και την παράγουμε εμείς, έχουμε την αλυσίδα παραγωγής. Αν αναπτυχθούν εκείνοι, θα πρέπει η παραγωγή να μεταφερθεί κατά ένα τμήμα της εκεί και να χαθεί από εμά. Αυτά τα πράγματα τα έχετε σκεφτεί, συμπεριλαμβάνονται με κάποιο τρόπο σε αυτές τις συμφωνίες, γιατί δεν τα βλέπω. Ούτε στις ΟΕΣ, ούτε στο TTIP, ούτε πουθενά. Αυτά και δεν ξέρω αν έχουμε υπολογίσει τι συνέπειες έχει αυτό σε άλλες περιοχές. Ευχαριστώ. Ο Σλάβος Κοράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα κυρία Επίτροπε και κυρία Γινάσου. Πιστεύω ότι ε, το TTIP ε, είναι μια συμφωνία που γεννήθηκε κάτω από ε, κακούς συνειρμούς και κακό αστέρι ε, γιατί πρόκειται στην ουσία για πολλές ε, μυστικές ε, συμφωνίες, διαπραγματεύσεις οι οποίες διόγκωσαν τη δυσπιστία. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, ε, υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου, κάποια μελέτη όσον αφορά την επίπτωση της συμφωνίας TTIP σε μικρές ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κυρίως στον Ειρηνικό και την Αφρική, πόσο μπορεί να διακινδυνεύσουν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης αναφέρθηκε, ελέγχθη, ότι ε, στις χώρες ΑΚΕ θα είναι πολύ μικρές ε, οι ε, οι επιπτώσεις, αλλά πολλές Ε, πολλές είναι οι μελέτες οι οποίες ε, λένε ότι θα ε, αυξηθεί κατά 1,7% περίπου η φτώχεια στις χώρες αυτές, ενώ αντίστοιχα η Κομισιόν λέει κατά 0,7% εάν και εφόσον. Το know-how των ε, ε, ε, τις ειδήσει προς τις χώρες της, της, των περιοχών ΑΚΕ μπορεί όμως να έχει αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά την, το land grabbing κλπ. Πιστεύετε ότι δεν πρέπει να προβλεφθεί τίποτα για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων ή προβλέπετε κάτι και δεν το γνωρίζουμε. Τελευταία ερώτηση αναφέρονται ε, ε, διάφορες ε, θετικές ας πούμε επιπτώσεις οικονομικές αλλά φαίνεται να διαφαίνονται και κάποιες κλιματικές και λοιπές ζημίες. Προβλέπετε κάτι στις μελέτες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτες. Und insofern finde ich es sehr spannend, diese Diskussion. Und Ich glaube, okay, κ. Σόλτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι ε, πολύ ε, σκόπιμο που κάνουμε μαζί την κοινή αυτή τη συνεδρία δύο επιτροπές. Το Ίδρυμά σας, κυρία Σβίκ, ξέρω ότι λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις με το TTIP προειδοποίησε για τις γεωπολιτικές αλλαγές. Θα γίνουν μεγάλες μετατοπίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, είχατε πει. Και τώρα που είμαστε σε μια προηγμένη φάση των διαπραγματεύσεων και για το TTIP και για άλλες συμφωνίες που ακούστηκαν προηγουμένως και με τον Καναδά, έχουμε φτάσει σε μια ε, ε, φάση που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε περί τίνο συζητούμε. Εάν πρόκειται για προδιαγραφές και πρότυπα και κανόνες, έχει πολύ μεγάλη σχέση ε, το να δούμε πώς θα ε, ε, διαμορφωθεί η μελλοντική παραγωγή. Γιατί για να κάνεις εμπόριο πρέπει να έχεις παράξει πρώτα. Άκουσα και τους τρεις πανελίστες και τους ευχαριστώ και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση προς όλους. Ε, στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής αξίας, τι γίνεται μεταξύ των διαφόρων οικονομιών που έχουν ας πούμε μία αντίστοιχη ανάπτυξη και χρονικά όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πάνε οι εταιρείε τους και πλασάρονται σε χώρες που ακόμα αναπτύσσονται. Δηλαδή αυτή η αλυσίδα παραγωγής αξίας και πλούτου πώς ρυθμίζεται και πώς επηρεάζεται με αυτές τις συμφωνίες. Στο εσωτερικό του TTIP δηλαδή, πώς ε, βλέπετε αυτή τη δυνατότητα και στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχει μια στοιχειώδης ανάπτυξη ώστε να καλύψουν το κενό και το έλλειμμα και να έχουν μια σωστή παραγωγή. Δεύτερη ερώτηση. Η Παγκόσμια Τράπεζα ήδη από το 2014 έχει αποδείξει ότι 50% ήδη ε, του ε, παγκοσμίου εμπορίου είναι εμπόριο μεταξύ χωρών νότου, νότου προς νότου. Κυρίως προϊόντα ε, είναι αυτά που συναλλάσσονται. Και μάλιστα έχουν και διαφορετική ανάπτυξη οι χώρες αυτές. Άρα, ερώτηση, αυτό το πρόβλημα πώς επηρεάζεται από τις διαπραγματεύσεις τη τυπική με τον Καναδά. Λαμβάνεται υπόψη, συμπεριλαμβάνεται εκεί. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια, γιατί η TTIP θα έχει μια μακροπρόθεσμη επιρροή με τελείως διαφορετικές πραγματικότητες, δημογραφικές, κοινωνιολογικές κτλ. Όταν η Αφρική θα έχει το 2040-2050 2,5 δισεκατομμύρια κατοίκους και η Ευρώπη 490.000, αν το προβάλλουμε, αυτό σημαίνει κάτι και τι σημαίνει. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται και με την εμπορική πολιτική για να επηρεάσουμε την ανάπτυξη. Σταματώ εδώ, θα μπορούσα να προσθέσω πολλά ακόμα, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση, πάρα πολύ συναρπαστική κλπ. Στο μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο αυτά το θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα δεν είναι εδώ. Ο Σέλφος Μποστινάρου θα είναι τελευταίος. Σας ευχαριστώ κύριε Συμπροέδρε. Κυρία Επιτροπέ, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και θα αναφερθώ στον Αντώνιο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο. Το 1998 είπε λοιπόν ότι η Αφρική σήμερα είναι η, το πρώτο θύμα της παγκοσμιοποίησης. Από τότε πολλά συνέβησαν, αλλά όχι απαραίτητα για καλό. Και ε, η Αφρική είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης ε, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην Αφρική. Η, το διεθνές εμπόριο θα μπορούσε να είναι τμήμα της απάντησης ε, στα προβλήματα που έχουμε και είναι πολλά στις σχέσεις μας με την Αφρική, διότι χωρίς ε, μία γενική, στρατηγική, ε, συνολική προσέγγιση στην Αφρική δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε άλλωστε και το πρόσφατα δημοσιευθέν κείμενο για την ε, μετανάστευση που αναφέρεται στην καλύτερη διακυβέρνηση, τεχνική ε, αρρωγή, ε, κατάρτιση, βοήθεια έτσι ώστε επιτόπου οι άνθρωποι καλύτερα να καταλάβουν τουλάχιστον τους κανόνες που επιβάλλουμε στην Αφρική. Δεύτερον, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον η Αφρική ε, θα έχει καλύτερη μεταπτυχιακή ικανότητα έτσι ώστε ε, να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το εισόδημα, να υπάρξει ανάπτυξη πραγματική έτσι ώστε οι πολίτες να είναι υποκείμενα της ανάπτυξης και όχι αντικείμενα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών γιατί με το παρόν σχήμα ή υπόδειγμα η Αφρική ε, ε, θα παραμείνει ε, περιοχή εξαγωγής πρώτων υλών, άρα δεν προχωράει με κανένα τρόπο. Δέστε λίγο την κρίση του έμπολα διαπιστώθηκε πλήρης αποτυχία, πλήρης ανικανότης αντιμετώπισης ε, του προβλήματος βάσει των στοιχειωδών ε, ε, δράσεων που οφείλει να αναλαμβάνει ένα στοιχειωδός λειτουργών κράτος. Πώς είναι δυνατόν από εκεί να φτάσουμε με μία μαγική μπαγκέτα στην ανάπτυξη. Εντάξει, με την TTIP λέμε θα υπάρξει, ε, ε θα αύξηση, αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος επενδυτής στην Αφρική είναι η Κίνα. Ε, ο πρώτος ε, εισαγωγέας πρώτων υλών από την Αφρική πάλι είναι η Κίνα. Και επομένως το TTIP, η συμφωνία TTIP δεν αφορά εμάς και την Κίνα, δεν είναι δηλαδή κάτι που διέπει εμάς και την Κίνα θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση έτσι ώστε να ληφθεί πραγματικά και σοβαρά υπόψη η Αφρική. Γιατί η Αφρική διορθώνω, γιατί η Κίνα θα εξακολουθήσει να έχει την ίδια στάση απέναντι στην Αφρική, άρα το ίδιο υπόδειγμα θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Τελειώνοντας να πω ότι η επόμενη μεγάλη μας πρόκληση όσον αφορά την μετανάστευση και όσον αφορά κυρίως την κλιματική μετανάστευση θα είναι η Αφρική. Κολέγκα. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Δεν έχουμε χρόνο λέει ο Πρόεδρος θα γίνει μια προσπάθεια απάντησης. Σας ζητώ να μην υπερβείτε τα πέντε λεπτά έκαστος. Θα ξεκινήσουμε με την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη γενικότερης συζήτησης ε, για την σχέση ε, και την ε, αμοιβαία ας πούμε λειτουργία της ανάπτυξης και του εμπορίου, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει σήμερα εδώ, αλλά βεβαίως οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να επανέλθω έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη γενική συζήτηση. TTIP. Γνωρίζω ότι ε, μερικοί αγαπάτε, άλλοι δεν αγαπάτε τη συμφωνία TTIP, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ε, συμφωνία η οποία διέπει τις σχέσεις της εμπορικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών και ουχή τις σχέσεις με την Αφρική. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαπραγματεύσεις σε 20, σε 20 διαφορετικά πλαίσια. Το TTIP είναι ένα από αυτά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε βεβαίω ότι μπορούμε να συζητήσουμε ποια επίπτωση μπορεί να έχει αυτή η συμφωνία σε τρίτε χώρε. Έχουμε κάνει μία πρώτη ε, έρευνα η οποία έχει δημοσιευθεί, μία δεύτερη η οποία θα δημοσιευθεί ω ονούπο και μία τρίτη η οποία θα δημοσιευθεί περί τα τέλη του έτου. Επίση, ε, σε πολλέ ε, χώρε μέλη έχουν συσταθεί think tanks τα οποία επίση θα δημοσιοποιήσουν τις, τα ευρήματά τους. Σε γενικές γραμμές πάντως όλες οι μελέτες ε, συγκλίνουν ε, στο συμπέρασμα ότι μικρή θα είναι η επίπτωση στις σχέσεις ε, με την Αφρική. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να λειτουργεί η συμφωνία TTIP, εάν θα χρειαστούμε κάποια μετριαστικά μέτρα. Ε, είναι γεγονός ότι το Δεκέμβριο θα προχωρήσουν ε, κάποια ε, πράγματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί στην, στο γύρο της Ντόχα και που αφορούν τις πιο φτωχές χώρες. Δεν θα αντιμετωπίσουμε βέβαια όλα τα προβλήματα, αλλά το βέβαιο είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε και κάποια παλιά προβλήματα της Ντόχα και κάποια καινούρια. Δουλεύουμε λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, δουλεύουμε επίσης με την έρμπα ας πούμε. Είναι κάτι που δεν έχει επιβληθεί από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες ή οτιδήποτε. Θα υπάρξουν κάποια προγράμματα που θα αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα για χώρες της Αφρικής. Διότι ναι, το εμπόριο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε ε, να σώσει τους ανθρώπους, να βγάλει τους ε, ε, ανθρώπους από τη φτώχεια. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμπόριο από μόνο του. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ε, και στο εσωτερικό των χωρών τεχνική βοήθεια, πολιτική στήριξη κτλ. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά στο, Aid for, στο πρόγραμμα Aid for Trade. Και ο μεγαλύτερο εταίρος βέβαια είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όταν μιλάμε για πρότυπα, ε, στο TTIP, στην TTIP έχουμε βάλει τεχνικά πρότυπα και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, τους ε, καλύτερους ε, επαγγελματίες θέσπισης προτύπων. Ας πούμε, εάν ε, δεχτούμε ότι ε, μπορεί ένα τεστ ε, για το κατά πόσον ένα χαλί είναι έφλεκτο, μπορούμε να δεχτούμε το τεστ το οποίο έχει γίνει στη μία πλευρά του Ατλαντικού, να το δεχτούμε και από την άλλη, γιατί να κάνουμε δεύτερο τεστ, γιατί να κάνουμε δεύτερη δοκιμή. Αυτά προσπαθούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας έτσι ώστε να γίνεται ένα τεστ και όχι δύο. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα. Πρότυπα ε, πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, της προώθησης της συνεταιριστικής ε, ευθύνης, που δεν θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους, αλλά οι χώρες θα κληθούν σε εθελούσια βάση να τις ε, σεβαστούν επίσης κάποιες ε, αρχές ε, για, την, για το σεβασμό προτύπων περιβαλλοντικών κτλ. Και πιστεύω ότι για αυτές τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν από πλευράς των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πιστεύω λέω ότι είναι θετικό να υπάρχουν κοινά πρότυπα και ότι αυτό θα είναι θετικό. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις βέβαια. Mm. Αλλά υπάρχουν και πολλέ οι οποίε δεν σχετίζονται με το σημερινό θέμα. Όπω σα είπα, κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαρίστω να επανέλθω οποτεδήποτε θελήσετε. Δεν δέχομαι δεν δέχομαι βέβαια τι αυτό που ακούστηκε ότι ε, η συμφωνία TTIP, ε, η διαπραγμάτευσή της έγινε ε, σε πλήρη αδιαφάνεια. Υπάρχουν εκατοντάδες σελίδες, πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι προσβάσιμες στο Κοινοβούλιο και και ε, στο, στους πολίτες και στο διαδίκτυο. Κύριε Κοράο, δεν, ε, οι εμπορικές συμφωνίες πάντα έχουν και ε, κάποια απόρριτα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, αυτά ήθελα να πω, θα σταματήσω εδώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για όλα αυτά που μας είπατε. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Γνάσουνου. Για πέντε λεπτά επίσης, παρακαλώ. Oui, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ε, φεύγουμε με κάποια, πώς να το πω, ανακούφιση ότι μας καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι. Μας το ξέραμε βέβαια από πριν, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται αυτό. Γενικώ, νομίζω, ξεκινάμε στραβά αν πούμε ευθύ εξ ότι δεν θα υπάρχει αρνητική επίπτωση από την TTIP για τις χώρες αυτές. Γιατί εάν δεν καταλάβουμε ότι ενδεχομένως υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, δεν θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι έχει σημασία να αναρωτηθούμε, να αλλάξουμε δυναμική και να ε, κάνουμε προβολές σε σχέση με τα όσα συμφωνήσαμε όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εάν δεν αλλάξουμε και δεν αναπτύξουμε τις οικονομίες των χωρών αυτών, ε, τότε ας αλλάξουμε θέμα και να ξεχάσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να κατεβάσουμε τα ρολά. Όταν η Ευρώπη υιοθετεί νέους κανόνες και ε, υπάρχει για τις χώρες ΑΚΕ μία ε, βοήθεια, μία συνοδεία και παρακολούθηση. Χρειάζονται χρόνο οι χώρες αυτές για να ευθυγραμμιστούν. Έχουμε ζήσει καταστάσεις τύπου Κένιας και αλλού όπου αρχίσαμε να εξάγουμε προϊόντα που είχαμε σταματήσει να εξάγουμε. Και δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί κανείς στους κανόνες αυτούς και να συμμορφωθεί γιατί οι λαοί ε, είναι οι πιο φτωχοί των φτωχών. Δηλαδή όταν του λες ότι το άλφα προϊόν που το παράγεις και το καταναλώνεις αιώνες ολόκληρους με αυτόν τον τρόπο τώρα πρέπει να αλλάξεις. Γίνεται, δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι υπάρχουν και δυνητικές αρνητικές συνέπειες. Ωραία. Ε, στο Κοτονού λοιπόν έχουμε αναλάβει κάποια δέσμευση όπου αμοιβαία αναγνωρίζουμε ότι η τάση είναι η απελευθέρωση, η φιλελευθεροποίηση και κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί. Πώς θα γίνει όμως να είναι αμοιβαία υποφελής και για τα δύο μέρη, δηλαδή και κυρίως για τις χώρες μας. Τίθε το ερώτημα, τη σωστή απάντηση δεν την έχουμε βρει ακόμα. Αυτό μας προβληματίζει. Πώς μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε για να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα παγκόσμια παραγωγής αξίας προς όφελος των κρατών μας. Πρώτη ευθύνη είναι δικιά μας. Στη γραμματεία ΑΚΕ προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, τις χώρες μας, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, για να μην μπούμε σε ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων γειτονικών και ομόρων κρατών και να έχουμε πραγματικές στρατηγικές. Όχι μόνο για τη δημιουργία ε, αλυσίδας ε, παραγωγής αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Εχθές το πρωί ήμουνα με κάποιον αιθίωπα παραγωγό και εξαγωγέα, που μου εξήγησε ότι είχε επιστρέψει από την Ιγυρία που τον είχαν καλέσει διότι εκεί ε, εισάγουν ντομάτα από την Ισπανία ενώ βγάζει και η Αιθιοπία ή και η ίδια η Νιγηρία και ε, το Μπορκίνα Φάσο. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να, να εισάγουμε πορτοκαλάδα από την Ισπανία, ενώ στο διπλανό χωράφι καλλιεργούν πορτοκάλια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε στήριξη, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εμείς ή άλλα μέσα αναπτυξιακά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συμμετέχουμε στη συζήτηση που γίνεται. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εκεί λίγο ανησυχώ οι διαπραγματεύσει TTIP δεν είναι αναπτυξιακέ, προφανώ και δεν είναι. Αλλά εάν οι δύο χώρε που το συζητάνε ήταν το ίδιο πρωταθλήτριε ε, το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, για να υπογράψουν τα δύο, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που συζητάνε μεταξύ τους έχουν επιπτώσεις και στους φτωχότερους των φτωχών. Εάν δεν προβληματίζονται, έχουμε μεγάλες δυσκολίες, δεν πρόκειται να τα βρούμε και να συνεργαστούμε. Ας ασχοληθούμε σοβαρά, να αρχίσουμε κατανοώντας το πρόβλημα, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα ε, όσο θα επιθυμούσαμε, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Έχουμε ενδεχομένως στη γραμματεία μας την ευκαιρία να υπάρχει μια νέα ομάδα που προχωράει προς μια νέα κατεύθυνση. Οι ΣΟΕΣ, ε, ε, συμφωνίες που υπογράφονται αυτό το καιρό, θα πρέπει να έχουν ευεργετικές επιδράσεις για τις χώρες. Αλλιώς θα παίζουμε το παιχνίδι των πολέμιων τους που είπαν ότι είναι τελείως άχρηστες. Αν ε, αδρανίσουμε θα δικαιωθούν εκείνοι και θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Σμίκ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σκέφτομαι τον κόσμο έτσι όπως είναι και δεν είναι ιδανικά πλασμένος. Έχουμε ένα, ένα πολυμερές σύστημα που δεν μεταξελίσσεται πάρα πολύ δυναμικά και έχει κάθε δικαίωμα εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάπτει διμερείς συμφωνίες. Και έχει και νόημα αυτό με το μεγαλύτερο εταιρικό, ε, εμπορικό εταίρο να κοιτάξουμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε από κοινού τις προϋποθέσεις για το εμπόριο. Εάν το καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις TTIP, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες μεν στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά αυτές δεν θα είναι τόσο δραματικές ε, τις επιπτώσεις τους για το λόγο που σας είπα. Και επίσης υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, να μειώσουμε ή να αποτρέψουμε τελείως αυτές τις συνέπειες. Τώρα, για τις ε, προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα τεχνικά, ε, και ε, στα θέματα υγείας και φυτοϊγειονομικής προστασίας. Αν βελτιωθούν τα στάνταρ θα έχουν προβλήματα οι αναπτυσσόμενες χώρες γιατί δεν έχουν ούτε τους θεσμούς, ούτε την ικανότητα, ούτε τις οικονομικές δυνατότητες να το αντιμετωπίσουν αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι αρκετά περίπλοκο και θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί στο βαθμό που δεν προχωρούμε σε προδιαγραφές για λόγους προστατευτισμού Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για προστασία των καταναλωτών, για την προστασία των εργαζομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα πρότυπα. Γι' αυτό και οι ίδιες οι χώρες οι αναπτυσσόμενες έχουν συμφέρον να ανέβουν τα πρότυπα και στην ίδια τη χώρα. Συχνά όταν προσπαθούν να αυξήσουν τα στάνταρ και τις προδιαγραφές οι αναπτυσσόμενες χώρες για να εξάγουν και προς εμάς, ταυτόχρονα προστατεύουν την υγεία και τους καταναλωτές τους δικούς τους. Οπότε έχει μεγάλη σημασία εκεί να δούμε τις ποιοτικέ υποδομές και να τις βελτιώσουμε. Αυτή είναι μια αφετηρία του Aid for Trade που είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, τα ιδιωτικά πρότυπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πέρα δηλαδή από τα νομοθετικά υποχρεωτικά και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήδη 80% ε, των γεωργικών εξαγωγών της Κένια ε, υπάκουαν σε εθελοντικές προδιαγραφές, πρότυπα που είχαν συμφωνήσει μεγάλες ας πούμε αλυσίδες ε, σούπερ μάρκετ για να μπορούν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που μπορεί να είναι ιδιωτικά, εθελοντικά, προαιρετικά και δεν θα πρέπει να είναι η απέτηση να κρατήσουμε και εμείς χαμηλά τα πρότυπα. Όχι, να ανεβούν τα δικά τους για να βοηθηθούν και χώρες αυτές ε, για τους ίδιους τους δικούς τους, επαναλαμβάνω, καταναλωτές και στην εχώρη αγορά. Για το θέμα των παγκοσμίων επιπτώσεων του TTIP και το ρόλο της Αφρικής. Είπα ότι φοβάμαι περιθωριοποίηση. Στο τέλος όμως της ομιλίας μου ανέφερα ότι υπάρχουν και άλλοι παραγόντες πολύ πιο σημαντικοί ε, που καθορίζουν για το τι κάνουν οι αφρικανικές χώρες αλλά και άλλες εμπορικές ροές ε, ειδικέ μας προς αυτούς. Ε, αναφέρθηκαν ορισμένοι τέτοιοι παράγοντες. Πώς αναπτύσσεται η Κίνα. Τι γίνεται με τη δημογραφική ανάπτυξη της Αφρικής. Θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050 ο πληθυσμός στην Αφρική. Εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι τελείως κομβικό αυτό το θέμα. Είναι τεράστια ευκαιρία. Το πρόβλημά μας στην Ευρώπη είναι ότι γυράσκει και ο πληθυσμός και οικονομικό πρόβλημα είναι και για τις επιχειρήσεις. Δεν βρίσκουμε ειδικευμένου εργαζόμενους. Αυτά όλα είναι πιο σημαντικά από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ήθελα να το πω όμως και το λέω. Η Ευρώπη έχει ευθύνη όταν ε, συνάπτει τέτοιες συμφωνίες να φροντίζει να περιορίζονται στο ελάχιστο τα αρνητικά και να ε, μεγιστοποιούνται τα θετικά. Μία μόνο παρατήρηση για το TTIP. Γιατί ε, συγκεντρώνει τέτοια προσοχή, γιατί θα είναι συμφωνία ελευθερών συναλλαγών μεταξύ δύο γιγάντων. Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες, αλλά ποτέ ε, δεν προκάλεσαν τέτοιο ενδιαφέρον στο παρελθόν. Πολλοί κόσμος φοβάται την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις της, που μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών. Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη. Κάποιος μίλησε για ανισότητα. Η ανισότητα είναι κάτι που ε, διαπιστώνουν πολλοί άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή, με τους φίλους, γνωστούς τους κτλ. Βλέπουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο παράγων εργασίας σε σύγκριση με τον παράγοντα κεφάλαιο έχει χάσει διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό δεν μπορεί ο κόσμος να το πει ε, με το όνομά του με οικονομικούς όρους, αλλά βλέπει τις συνέπειες γιατί τις υφίσταται. Και η πολιτική περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Τα είπε και η κυρία Μάλμστον. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν, δεν μπορούμε να αναμένουμε εμπορική πολιτική, μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα και θα δώσει τις λύσεις. Ε, αυτό που έχει σημασία και ανέφερα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα συνολικό πακέτο με στόχους, λένε ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα λυθούν. Και η εμπορική πολιτική ε, θέλει προσοχή για πολλά σημεία, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα όλα, ή να εξασφαλίσει τον, το μέλλον μας. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για να ξέρουμε κάπως που κινεί τη συζήτηση και σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την παρέμβασή σα Στάνουμε, έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την πολύ πλούσια και πυκνή συζήτηση. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την ε, συνεδρία, θα ζητήσω στον συνάδελφο Λάγκε να κλείσει την συνεδρία σε αυτή. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεσίλια Μάλστρομ, την ε, Επίτροπό μα για το εμπόριο και τον κύριο Κινάσου από την ε, γραμματεία ΑΚΕ και τη Β' ΣΜΙΚ από το Ινστιτούτο που εκπροσωπεί για τις σημαντικές προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις θα τις ε, συζητήσουμε και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και θα τις λάβουμε υπόψη στις ε, συζητήσεις που κάνουμε για το TTIP. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω και δύο πιο γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτό που πετύχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως διαφάνεια δεν θα πρέπει να το αμφισβητούμε. Έχουμε πετύχει το να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του TTIP και οι 751 βουλευτές του Κοινοβουλίου και στις διαπραγματεύσεις να ε, βγαίνουν όλες οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο και όλα τα πρακτικά των διαπραγματευτικών γύρων. Τόση διαφάνεια πια δεν την έχει δει κανείς ποτέ και είναι και υποδειγματική και παράδειγμα προς μίμηση και θα πρέπει να το αξιολογούμε ως κατάκτηση του Κοινοβουλίου και να μην ε, βγάζουμε περσινά ξινά στα φίλια κάθε φορά. Επίσης, θα πρέπει να συζητάμε και να ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, να επιτύχει και τι δεν μπορεί να πετύχει μια ε, εμπορική συμφωνία και από πλευράς οικονομικής, ε, κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Υπάρχει ένα ζήτημα συνέχειας και συνέπειας των πολιτικών μας. Δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα της αναδιανομής του πλούτου και της ανισότητας ε, ή τα περιβαλλοντικά με μια εμπορική συμφωνία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ισχύει και για το TTIP και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ότι αυτό που μπορεί να θεωρείται απειλή, ακούσαμε, ε, μπορεί να αλλάξουν, ε, ε, να μετατοπιστούν κάποιοι τρόποι εμπορίου και κάποιες παρακάμψεις να γίνουν. Ακούσαμε για την περιθωροποίηση ενδεχομένως κάποιων χωρών. Αυτό στις διαπραγματεύσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες που μπορούμε να δράξουμε. Παράδειγμα, αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων και προδιαγραφών και για τρίτες χώρες. Και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό με τα πρότυπα και τον καθορισμό τους, πώς να το πω, με βρίσκει με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια ακούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στις προδιαγραφές μας και για το TTIP θα πρέπει να παραμένουν πολύ ψηλά και σήμερα έχω την εντύπωση ότι καλά δεν πειράζει να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας γιατί έτσι θα έχουν καλύτερη πρόσβαση κάποιες τρίτες χώρες. Ε, δεν γίνεται έτσι όμως πώς θα πάει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμβιβασμούς και εκδόσεις όταν πρόκειται για τεχνικές προδιαγραφές και για τρόφιμα. Θα τα καλύτερα για τον κόσμο όλα αυτά. Ε, στις διαπραγματεύσεις του ΤΙΤΕΠΗ e να ανοίξουν για τις τρίτες χώρες χωρίς εκπτώσεις όμως να τα τηρούν και να μπορούν να τα πληρούν όλα αυτά. Ας πούμε το Aid for Trade και υποστήριξη της δυνατότητας και της, και της ε, οικοδόμησης δυνατοτήτων μάλλον των χωρών αυτών. Όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε και αύριο για τη ρυθμιστική συνεργασία, κανονιστική συνεργασία για τα πρότυπα και για τις τρίτες χώρες. Κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό είναι τέτοιες περιφερειακές συμφωνίες πάντα να εντάσσονται στα πλαίσια του ΠΟΕ και όχι να απεμπολούμε τον ΠΟΕ, απλώς είναι συμπληρωματικά. Έτσι ώστε τελικά να έχουμε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας και να έχουμε παγκόσμιες όντως αλυσίδες παραγωγής ε, πλούτου και αξίας. Αυτά. Οπότε σήμερα δεν μπορούμε να πούμε αν είναι καλό ή κακό το TTIP για τις αναπτυσσόμενες χώρες ακόμα. Αυτό που έχει σημασία είναι τα κρίσιμα στοιχεία που συζητήσαμε να ληφθούν υπόψη και να διαμορφωθεί η συμφωνία έτσι ώστε να μην είναι κακή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό θα το λάβει υπόψη του στη συζητήση στο σύνολο της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια έχω να πω κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να φύγουμε με παρεξηγημένοι. Εγώ ο ίδιος μίλησα για στάνταρ και τον αντίκτυπο. Είμαι υπέρ της σύγκλησης των ε, κανόνων των προδιαγραφών ποιότητας προς τα πάνω. Αναφίβολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα μπορούν να ανταποκριθούν οι χώρε ε, οι αναπτυσσόμενε. Ε, η απόψη μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ορίσουμε μια στρατηγική που θα επιτρέψει στι αναπτυσσόμενε χώρε να προσαρμοστούν σε αυτού του ρυθμού προ τα πάνω. Γιατί διαφορετικά έχουμε πρόβλημα. Και εδώ περιμένω από την Κομισιόν μια, ένα ανακοινοθέν που θα ξεπερνά αυτέ τι πτυχέ που μα παρουσίασε η κυρία Μάλστρομ, που προσπάθησε να συμπεριλάβει τις επιθυμίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Αλλά αυτή η στρατηγική πρέπει να ε, τελειοποιηθεί. Και ο κύριος ε, Νασανού προς αυτή την κατεύθυνση μίλησε. Έχουμε μία, ένα προβληματισμό. Πρέπει αυτό να το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Σάρλα. Μπορούμε να συζητήσουμε να συνεχίσουμε διμερώς τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους μας που είναι σήμερα εδώ. Μας μένουν δύο σημεία στην ημερήσια μας διάταξη που πρέπει να τα ολοκληρώσουμε. Για τα διάφορα έχουμε το σημείο 17. Έχουμε εδώ ερω... στα διάφορα κάτι. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas de questions, Εάν δεν έχετε θέματα στα διάφορα, να μιλήσουμε για το τελευταίο θέμα που είναι η ημερομηνία της ε, διεξαγωγής επόμενης μας συνεδρίασης. Είναι ε, τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 από τις 3 μέχρι τις 6 και 30 το απόγευμα και την Τρίτη 9 με 12.30 και 3 με 6.30 11 και 12 Ιουλίου Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και εδώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για σήμερα. Θα ακολουθήσει η, συνάντηση, η συνεδρίαση των συντονιστών και ζητώ από όσου δεν είναι συντονιστές να εγκαταλείψουν την αίθουσα σιωπηρό, ώστε να μπορέσουμε οι υπόλοιποι να συνεδριάσουμε. Donc, euh, ceux qui ne sont pas concernés, quittez la salle en silence et le plus vite possible, s'il vous plaît. Quant à moi, je vais céder ma place à notre collègue Nir Deba, qui va présider la. Ο κύριος Δέβα θα προεδρεύσει συνεδρίαση των συντονιστών. Είμαι υποχρεωμένος να, να φύγω. Του δίνω και το λόγο και τη θέση του Πρόεδρου.